Διατλαντικό εμπόριο και σχετικές ε, σχέσεις επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα σε ό,τι αφορά τι δημόσιες συμβάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς φορείς. Καλώς ορίσατε λοιπόν και καλώς ορίζουμε και τους πανελίστες που μας ακούν και ήλθαν εδώ και οι διαπραγματεύσεις για το TTIP είναι ε, ουσιώδους σημασίας για την ε, Επιτροπή μας ε, και σε θέματα υποποίησης και σε θέματα δημοσίων συμβάσεων που θα συζητήσουμε σήμερα. Έγινε πριν μια πρώτη κοινή συνάντηση μεταξύ μου και του κυρίου Λάγκε το Φεβρουάριο πέρσι. Εξετάσαμε τα πρότυπα σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές και είπαμε ότι τα θέματα δημοσίων συμβάσεων ε, θα τα κάναμε πιο μετά και αυτό λοιπόν ε, καλούμαστε να κάνουμε σήμερα. Έχουμε συνεργασία σε ό,τι αφορά κυρίως τα οχήματα και άλλα θέματα μεταξύ των οποίων και η προστασία των καταναλωτών. Θα προεδρεύσω του πρώτου τμήματος ε, της ακρόασης και ο κύριος Λάγκε θα προεδρεύσει του δεύτερου της τμήματος. Ο κύριος Λάγκε να πάρει το λόγο, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φόρτα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, τώρα άνοιξε το μικρόφωνο του. Ο πρόεδρος τον ευχαριστούμε. Κυρία Πρόεδρε Φόρτ, Αγαπητοί συνάδελφοι, όντω το θέμα των δημοσίων συμβάσεων σε ό,τι αφορά τη διαπραγματεύση στη ΤΥΠ είναι, θεωρώ, ίσω το κατεξοχήν ε, κρίσιμο ζήτημα. Και εμεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε ό,τι αφορά την αγορά δημοσίων συμβάσεων τη ΕΕΠΑ. Ξέρω ότι είναι 12% του ΑΕΠ τη αγορά στις ΕΕΠΑ. Και ξέρετε ότι στη ΣΥΠΑ διάφορα ζητήματα εξαιρούνται τον, του, του κλάδου των δημοσίων προμηθειών σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίκαιρη πολύ αυτή η συζήτηση, γιατί την Κυριακή ο πρόεδρος ε, Ομπάμα θα επισκεφθεί ε, το Ανόβερο και ενδεχομένω να παρουσιάσει, να κάνει δηλώσεις οι οποίες θα δώσουν νέα ορμή νέα ταχύτητα στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν κατά τη τελματώσει στην ε, παρούσα φάση. Θα ήταν λοιπόν αυτό απαραίτητο αν θέλουμε όντω να πετύχουμε τη συμφωνία αυτή και μάλιστα υπό την κυβέρνηση Ομπάμα. Κρίσιμη φάση λοιπόν στις διαπραγματεύσεις και ως εκ τούτου Είναι πραγματικά πολύ επίκαιρη η σημερινή ανταλλαγή απόψεων για θέματα δημοσίων συμβάσεων. Στο πρώτο τμήμα της ε, ακρόασης θα προεδρεύσει η συνάδελφος πρόεδρος ε, κυρία Φόρτ σε ό,τι αφορά την εσωτερική διάσταση των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δεύτερο τμήμα θα προεδρεύσω εγώ και θα ασχοληθούμε πιο πολύ με το ζήτημα του πώς διεξαγάγονται οι διαπραγματεύσεις και τι δυνατότητες έχουμε να προσχωρήσουμε στην αγορά δημοσίων συμβάσεων των ΕΠΑ. Και μάλιστα με ένα διαφανή και συγκεκριμένο τρόπο. Είμαστε έτοιμοι νομίζω και οι εκπρόσωποι μας είναι εδώ. Η ατζέντα είναι σαφώς ορισμένη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, Πρόεδρε. Μάλιστα, ο κύριος Φίλιπ Σίτρον, Στρέν, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του European Rail Industry. Μετά έχουμε την κυρία Τζιν Σεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πλοίων και Ναυτιλιακών Εξοπλισμών και τον κύριο Ντάνιελ Μπάσο τέλος από την ΕΤΟΚ, την Ομοσπονδία ε, εργαζομένων. Θα δώσουμε λοιπόν πέντε λεπτά στον καθένα. Α πάρει το λόγο ο πρώτο ομιλητή, ο κύριο Φιλίπ Σίτροεν. Merci Madame le Président. Merci aux deux comités et INTA de m'avoir invité. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις δύο επιτροπέ για την πρόσκληση. Έχω προετοιμάσει τις διαφάνειες μου στα αγγλικά, αλλά η παρουσίαση μου θα γίνεται στα γαλλικά. Mm-hmm. Έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε και από τις δύο πήγε. Εγώ δεν βλέπω τι διαφανίες μου και ωρα. Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα εγώ να ξεκινήσω να λέω είναι ότι η διαπραγμάτευση για την τύπη για εμά είναι εξαιρετικά σημαντική. Η... Μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Γιατί πολλές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στην Ένωσή μας, στην UNIFE, ε, δραστηριοποιούνται στην Αμερικανική αγορά. Ωστόσο, όπως βλέπετε σε αυτήν την διαφάνεια, έχουμε το 84% της αγοράς, ε, το μερίδιο της αγοράς στην Ευρώπη, ενώ το 46% μονάχα παγκοσμίω. Στην διαφάνεια που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σας βρίσκεται τα λογότυπα όλων των εταιριών μελών της UNIFE που δραστηριοποιούνται ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε την εξέλιξη της αγοράς. Ε, περιμένουμε μια αύξηση κατά 3,3% της ε, ζήτησης, φτάνοντας σε, στο ύψος των 22 δισεκατομμυρίων ε, δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για εμάς και Εξ όσων γνωρίζω, ε, προετοιμάζεται και μια έκθεση μια συμβουλευτική ε, εταιρεία για την εξέλιξη της Αμερικανική αγοράς. Εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, με τη συμφόρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα μια αγορά μεταφοράς φορτίων που αναπτύσσεται. Υπάρχουν ορισμένε ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πολλά προβλήματα παραμένουν όσον αφορά την πρόσβασή μα. Τα κυριότερα είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα οι περιορισμοί που θέτουν οι, ε, τα όρια δεσμεύσει για τις δημόσιε συμβάσεις που θέτουν ε, το καθεστώ του ΠΟΕ, ε, το οποίο καλύπτει 37 πολιτείε των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίση, στο ομοσπονδιακό επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει η, το Buy America Act, μια νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι το 60% του τροχαίου του υλικού πρέπει να αγοράζεται από αμερικανικές εταιρείε. Και ε, όσον αφορά τις, τις, ε, τους σιδηροδρόμους τους ομοσπονδιακούς εκεί το ποσοστό είναι 100% πια. Σε συγκεκριμένες πολιτείες μάλιστα υπάρχουν και πιο συγκεκριμένοι νόμοι όπως για παράδειγμα στην Καλιφόρνια οι τάση στον τομέα των σιδηροδρόμων διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έντονη πολιτική πίεση να αυξηθεί η χρήση υλικού παραγωγόμενου στι στις ΗΠΑ στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Κάτι σημαντικό πρέπει να γνωρίζετε. Το τέλος 2015 το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε ένα πρόγραμμα 305 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πέντε χρόνια επενδύσεων, όχι μόνο στους σιδηροδρόμους, αλλά και αλλού, Fixing America Surface Transportation Act, γενικώ για τις επίγειες μεταφορές. το οποίο προβλέπει μια ανάπτυξη της τάξης του 10% μέχρι το οικονομικά του 2020. και το ποσοστό του 60% που σας ανέφερα προηγουμένως θα ανέβει στο, 10, στο 70% μέχρι το 2020, το οποίο <clears throat> δεν μας ευνοεί εμάς, τις, ευρωπαϊκέ τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Χρησιμοποιείται επίσης, μάλλον σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στη Βοστόνη, ε, και πάλι υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και να προτιμάται το παραγόμενο στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει τη σύνταξη νομοθεσία, η οποία θα μπορούσε να ε, θέσει περιορισμούς στις προσλήψει του προσωπικού να προτιμώνται εργαζόμενοι τοπικά όταν τα έργα χρηματοδοτούνται από ομοσπονδιακά κονδύλια. Ποιε είναι οι κυριότερε ανησυχίε ε, ε, των ευρωπαϊκών κατασκευαστών τροχαίου υλικού. Όλα αυτά που σα είπα έω τώρα ε, δείχνουν ότι αυξάνονται οι προϋποθέσεις από το, στο επίπεδο των πολιτιών και στο ομοσπονδιακό επίπεδο που ζητούνται το υλικό να έχει, κατασκευαστεί το, τοπικά. Επίσης θεωρούμε ότι οι, οι περιορισμοί στις προσλήψεις που τίθενται και αυτοί δεν μπορούν να ε, λειτουργήσουν σε βάθος χρόνου και ταυτόχρονα σε διάφορες πολιτείες αυξάνονται οι συγκεκριμένες ειδικέ τους προς την πολιτεία απαιτήσει. Τα συμβόλαια, για παράδειγμα, στο Σικάγο και τη Βοστόνη πλέον έχουν ε, τα κέρδισαν ε, κινέζικες εταιρείες μετά από συγχώνευση. Ποια είναι λοιπόν τα μηνύματα που θέλει να σας περάσει η ένωσή μας, η UNIFE. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια ενιαία αγορά μεταξύ Ευρω... Ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ όσον αφορά τους σιδηροδρόμους ε, χωρίς τερμπλώσεις του ανταγωνισμού οι περιορισμοί που θέτουν οι ΗΠΑ καλύπτουν και, τις ομοσπονδιακές, και τα ομοσπονδιακά συμβόλαια, αλλά όλο και περισσότερο πολιτείες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πολιτική που ακολουθεί η Αμερικανική κυβέρνηση όσον αφορά τι δημόσιε προμήθειε θα πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οποιασδήποτε πρωτοβουλίε για προώθηση τη απασχόληση σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να, να μην αφορούν ε, τους, ε, την κα, κατασκευή σιδηροδρόμων, κατά την άποψή μα. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Γνωρίζουμε την, πόσο ευαίσθητη είναι η διαπραγμάτευση και βλέπετε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ευαίσθητη όσον αφορά τα, που θεωρούνται αυτά τα θέματα ευαίσθητα στις ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Σέν θα μας μιλήσει για την αυτιλία. I'm the trade policy advisor at... Jim Sen γίνομαι και είμαι σύμβουλος πολιτικής ε, στο C Europe. Οπότε θα, πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται με του, αυτούς που ναυπηγούν τα πλοία δεν είναι ούτε πλειοκτήτες ούτε φοβιστές είμαστε επομένω 100% εκπρόσωποι της, του συνόλου ε, της ε, ναυπηγής 91 δις είναι ο τζίρος του και 500.000 ε, θέσεις απασχόλησης και 400.000 έμεσα είναι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούμε. Το, το C-Europe έχει αναπτύξει ε, μια αξιόλη δραστηριότητα όσον αφορά θέματα του TTIP και στείλαμε στην Washington κάποια αντιπροσωπεία για τα εμπορικά θέματα να μιλήσουμε με τους εμπλεκόμενους Αμερικανούς και πήγαμε διότι έχουμε διάφορους περιορισμούς όσον αφορά την ναυτιλία και έτσι υπάρχει πρόβλημα στο ε, να απολύσουμε τα πλοία που ναυπηγούμε στην Αμερική. Επομένως, έχουμε τους περιορισμούς ε, για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά υπάρχει και ένας νόμος να σας, που λέγεται Jones Act είναι ένας νόμος ένας νόμος 100 ετών και απαιτεί μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων να γίνει μεταξύ δύο σημείων στην Αμερική από αμερικανικό πλοίο με αμερικανικό πλοίο και από αμερικανική σημαία. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Οπότε δεν μπορούμε με ευρωπαϊκά πλοία να κάνουμε ε, τέτοιου είδους μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β στις ιπα ε, Μπορούμε να τα πάμε μέχρι την Αμερική, αλλά όχι ε, να κυκλοφορήσουμε και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Οπότε να δούμε ε, ακόμα και μέσω του TTIP αν λυθεί μέσω το πρόβλημα παραμένει το πρόβλημα ακόμα και αν ε, δεν έχουμε τον νόμο αυτόν στα πόδια μας έχουμε τις, ε, τους περιορισμούς που επιβάλλονται για τις δημόσιες συμβάσεις εδώ μπορεί να δείτε ορισμένα παραδείγματα κάποιων εξειδικευμένων σκαφών υψηλής τεχνολογίας που είναι ευρωπαϊκά αλλά καλύπτονται από τους κανόνες αυτών των περιορισμών προμηθειών που είπαμε και ακριβώς λόγω αυτού του νομοθετήματος δεν μπορεί ποτέ αυτά τα σκάφη να μπουν στην αγορά των ΙΠΑ το οποίο αποτελεί για εμάς ένα πρόβλημα. Επίσης είναι πρόβλημα και για τους Αμερικανούς. Γιατί, διότι, να, κοιτάξτε τα παγωθραυστικά ως παράδειγμα. Είναι ισχυρή, μεγάλη χώρα οι ΗΠΑ, αλλά Η ειρωνία είναι ότι έχουν μόνο δύο παγωθραυστικά τα οποία είναι και αρκετά παλιά, 40 ετών και μόνο ένα από τα δύο λειτουργεί. Το άλλο παγωθραυστικό έχει κάνει βαλιστή ούτως ώστε να συντηρηθεί το άλλο. Γελία κατάσταση. Οπότε για να μπορέσουν να καλύψουν το έδαφος ε, ως προς τους ε, ε, Ρώσους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην Αρκτική, είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, θα πρέπει να βαθμίσουμε το στόλο μας. Οπότε θα πρέπει να φυγήσουμε τρία μεγάλα παγωδραστικά. Όμως το πρόβλημα με τη ΣΥΠΑ είναι ότι για να αναφυγήσουν εκεί ένα παγωδραστικό χρειάζονται ένα δι ε, δολάρια και θα τους πάρει 10 χρόνια να τον αναφυγήσουν Αλλά εκτό από αυτό δεν έχουν τεχνολογία. Πρέπει να την αγοράσουν από την Ευρώπη. Και ακόμα και αν λύσουν αυτά τα προβλήματα αν βρούνε το ναυπηγείο, βρουν την τεχνολογία και τα χρήματα, θα έχουν ακόμη πρόβλημα, διότι το νέο σκάφος ποτέ δεν θα είναι έτοιμο ε, πριν το παλαιό παγοθραυστικό κλείσει τον κύκλο ζωής του. Αυτό είναι πρόβλημα, πρέπει να ανέβουν μια λύση και να η λύση εδώ ή στην Ευρώπη. Διότι, όπως σας είπα, ε, έχουμε την τεχνολογία και την εμπειρία. Και επίσης η τιμή που ζητούμε είναι το 1 τρίτον της Αμερικανικής και επίσης θα παραδώσουμε το σκάφος σε πολύ συντομότερο χρόνο. Αλλά παρά το TTIP, λόγω των περιορισμών, δεν μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, τα πλοία μας. Οπότε ε, βλέπετε ποιες είναι οι σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά και τον εξοπλισμό των πλοίων. Γιατί υπάρχει ένα άλλο νόμο που λέει ότι θα πρέπει κατά 60% ε, το, τα, το, ο εξοπλισμό να είναι ε, από ντόπια προϊόντα. Άρα δεν είναι δυνατόν ε, να, προχωρήσουμε να προχωρήσουμε με αυτό το νόμο και αυτά τα πλοία που καθαρίζουν τα λιμάνια αυτή η βυθοκόρη δεν είναι δυνατόν να ε, λειτουργήσουν γιατί είναι βαριά πλοία γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με το, αυτό το 60 και 40% ε, λόγω ακριβώς αυτής της, του περιορισμού του 60% ντόπιου εξοπλισμού. Επόμενη διαφάνεια. Και με όλον αυτόν τον προστατευτισμό και αυτούς τους περιορισμούς τελικά τι έγινε. Δεν υπάρχει πλέον ε, ναυπηγική. Ενώ εδώ ακμάζει ναυπηγική και είμαστε πρωτοπόροι στην παγκοσμία αγορά. Πιστεύουμε στην ε, ελεύθερη αγορά και βρίσκουμε θέσεις στην αγορά για τα προϊόντα μας. Βλέπετε ότι έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Αλλά βέβαια υπάρχει πάρα πολύ αθέμητο συναγωνισμό στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίω στην Αποανατολή, γιατί έχουμε παράνομε κρατικέ παρεμβάσει, έχουμε ε, προκαθορισμό παράνομα χαμηλών τιμών και άρα δεν ισχύουν ε, οι δίκαιοι κανόνε ε, του παιχνιδιού εκεί. Οπότε, η θέλω να σα πω το μήνυμά μα που είναι απλό. Εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορέσουν να ανοίξουν την αγορά των ε, προμηθειών όσον αφορά ε, την ναυπική και την ε, αγορά μας αυτή στην Ευρώπη. Εμείς μπορούμε να τους ναυπηγήσουμε όλα τα πλοία, όσα, όλα όσα χρειάζονται. Πρόεδρος. Ε, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Όποιος θέλει αυτές τις μπορεί να τις βρει στο website της Επιτροπής μας κάποια στιγμή αργότερα γιατί κάποια σημεία Πρέπει να τα ξαναμελετήσουμε. Ο τρίτος μιλής είναι ο Ντανιέλ Μπάσο από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Και μετά θα σημειώνουμε και ποιο θέλει να πάρει το λόγο στο κατάλογο των ομιλητών, λέει η Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Ντανιέλ Μπάσο θα επικεντρωθώ πιο πολύ στην ευρωπαϊκή πλευρά και όχι τόσο στην αμερικανική. Κατανοούμε το θέμα αυτό. Α, ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι υπάρχει συμφέρον αμυντικό προς τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Και συνεργαζόμαστε με τους, Αμερικανικούς, ομολόγου μα ομολόγους μας και τους Καναδούς ομολόγους μας σε ό,τι αφορά την Συμφωνία ΣΥΤΑ και τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ε, Δημοσίων Υπηρεσιών Θεωρούμε ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει ως σκοπό να έχει τη μείωση της ανεργίας, ε, να προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη και να δίνει απαντήσεις στις τοπικές ε, ανάγκες των Δήμων και των κοινοτήτων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι στην Ευρώπη το ίμιση των δημοσίων προμηθειών λαμβάνει χώρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι οι συνδικαλιστές ε, στην, Αμερική, Αμερική είναι ένθερμοι υποστηρικτές ε, της, ε, της νομοθετικής πράξης για να αγοράζουν μόνο αμερικανικά προϊόντα, το Buy American Act. Και υπάρχουν φυσικά και αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έχουμε δύο σημεία ο σημεία αφετηρίας. Καταρχάς, η σύμβαση του ΆΕΛΟ της, Ευρωπα... της ε, Παγκόσμιας ε, Οργάνωσης Εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις και κατά δεύτερον έχουμε και την Ευρωπαϊκή ε, Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Προφανώς τα δύο αυτά νομοθετήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, δεν θέλουμε να υπονομευθούν ούτε από την DTIP, ούτε από τη ΣΥΤΑ, ούτε από οποιαδήποτε άλλη μετέπειτα εμπορική σύμβαση. Γιατί την συνθήκη του 1994 τώρα, του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Είναι παλιά. Αλλά περιλαμβάνει σημαντικές ε, διατάξεις σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες και προβλέπει και κυρώσεις αν αντιρρηθούν αυτές οι προδιαγραφές. Επίσης προβλέπει την εφαρμογή των τοπικών συμφωνιών. Ωστόσο, δεν έχει επικυρωθεί αυτή η συνθήκη ούτε από τη ΣΥΠΑ, ούτε από τον Καναδά και μόνο από 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επικυρωθεί. Καλούμε λοιπόν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη το συντομότερο δυνατόν να επικυρώσουν την σύμβαση αυτή, τη συνθήκη αυτή. Εν συντομία τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, θεωρούμε ότι μας ικανοποιεί γιατί ε, προβλέπει θετικά στοιχεία και μια δεσμευτική κοινωνική ρήτρα μεταξύ άλλων που περιλαμβάνει βασικά αιτήματα των συνδικάτων, όπως για παράδειγμα απαιτήσει για τις συλλογικέ συμβάσεις, κοινωνικά κριτήρια, μεγαλύτερη διαφάνεια. Μας ικανοποιεί ως εκ τούτου η οδηγία αυτή. Η οδηγία αυτή το 2011 πέρασε αποφάση αναθεώρηση. Ξεκίνησε μάλλον η αναθεώρηση όπως θα θυμάστε. Και ήταν ευνοϊκή τότε η πολιτική κατάσταση, αλλά ε, και μάλλον ε, καταφέραμε να κάνουμε τη φωνή μας ακουστή, να ακουστεί. Έγιναν διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών μελών, κοινοβουλίου, το, της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Το 2004 πέρασε η οδηγία και έπρεπε να έχει εφαρμοστεί μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Άρα, χαιρόμαστε ε, που υπάρχει αυτή η οδηγία και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να υπονομευτεί από το TTIP. Επίση, αναγνωρίστηκε στην οδηγία η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Πολύ σημαντικό αυτό για μα. Και η σημασία των κοινωνικονομικών φορέων ε, και των παρόχων τέτοιων υπηρεσιών. Επίσης, μειώθηκε σημαντικά το κριτήριο του χαμηλότερου κόστους συμπερασματικά τα κινήματα συνδικάτων δεν θέλουν να θεωρηθούν στις δημόσιες συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις και το κόστος ως ε, ε, μη δασμολογικό εμπόδιο και θα θέλαμε αυτοί οι μηχανισμοί να λεφθούν υπόψη. Να υπενθυμίσουμε δε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εμπορικές συμφωνίες ε, δέχονται και σέβονται τα πρότυπα αυτά και επίσης οι ρήτρες δημοσίων συμβάσεων θα συνάδουν με το δεύτερο γενές δίκαιο για να μην υπάρχει οποιαδήποτε σύγχυση και αντίφαση μεταξύ του ευρωπαϊκού δικαίου και των τοπικών ε, προδιαγραφών αλλά και των ε, μεγάλων εμπορικών συμφωνιών. Και στο σημείο αυτό θα σταματήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Στην παρούσα φάση, λέει η πρόεδρο έχουμε 20 λεπτά που προβλέπονται για τις απαντήσει. Τέσσερα άτομα μόνο μου έχουν ζητήσει το λόγο. κυρία Γκραπίνη, η κυρία Ρένα, Ντάντον και η κυρία Γκέπχαρτ. Άλλος, κανείς, θέλει το λόγο. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την συζήτηση σε ό,τι αφορά το TTIP, σε ό,τι αφορά το θέμα των δημοσίων προμηθειών. Σας έλεγα ότι σας συγχαίρω που είχατε την ιδέα αυτή για να διοργανώσετε τη συζήτηση αυτή. Να ευχαριστήσω δε και όλους τους πανελίστες για τις παρουσιάσεις τους που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δυστυχώς θα πρέπει να πω ότι κάπως ε, Εκπλήξομαι και ενίσταμαι με αυτά που ακούω. Εγώ ε, το προηγούμενο έτος οργάνωσα μία παρόμοια ακρόαση στη χώρα μου και θα πρέπει να σας πω ότι σκύψαμε στα ίδια θέματα. Ευχαριστώ με τον κύριο Λάνε, που έθεσε το θέμα αυτό εκ νέου σήμερα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πω ότι εντοπίζω δύο μεγάλα προβλήματα. Η συνδρομική βιομηχανία καθώς και η ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτές οι δύο βιομηχανίες, αυτοί οι δύο κλάδοι πλήττονται από αυτά που συμβαίνουν σήμερα και φυσικά εξαρτώνται πάρα πολύ από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό το έχουμε υπόψη μας. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ τη εναρμόνιση των προτύπων, των προδιαγραφών και το του ανοίγματο τη αγορά. Γιατί στην Ευρώπη, ξέρετε, δεν έχουμε αντίστοιχο νομοσχέδιο με το Buy American, το American, Buy American Act για να προτιμούμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Έτσι λοιπόν η κατάσταση δεν θα είναι ακριβώς η ίδια για μας στην Αμερική και δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να ασκήσει πίεση επί των διαπραγματευτών που έχουν ε, πάρει εντολή από εμά να διεξαγάγουν τι διαπραγματεύσει για να υπάρχει ισορροπία σε ό,τι αφορά την πώληση προϊόντων, την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, γιατί διαφορετικά ε, θα βρεθούμε σε δυσχερή θέση στην Ευρώπη, σε μειονεκτική θέση. και θεωρώ ότι υπονομεύονται και τα πρότυπα προστασία των καταναλωτών. Γνωρίζουμε ποια είναι τα πρότυπα ε, στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα θέματα. Η Ευρώπη έχει νομοθετήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά ε, το ζήτημα αυτό, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, ε, την προστασία του καταναλωτή, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στην, στην Αμερική. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε λοιπόν την πίεση αυτή ε, στους ε, διαπραγματευτές μας από πλευρά της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Sorry Κυρία Ρένα, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Το όνομα Μαρία δεν είναι και τόσο σπάνιο. Υπάρχουν πολλέ σα που ονομάζονται Μαρία, επομένω λογικό να μπερδευτείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του δύο μελητέ και οι δύο παρουσιάσει ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Ε, σταθήκαμε στον τομέα των δημοσίων προμηθειών και οι ναυπηγικοί και οι σιδηρόδρομοι έχουν τη σημασία τους. Εγώ έχω τις εξής ερωτήσεις. Η πρόσβαση στην ε, αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται ότι θα πρέπει να είναι για εμάς μια κόκκινη γραμμή για να αποδεχθούμε την TTP όχι, δηλαδή κάτι το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να κερδίσουμε για να ε, αποδεχθούμε ε, την TTIP. Αναγνωρίζω ότι είναι κάτι σημαντικό να τεθεί στις διαπραγματεύσεις. Αλλά αναγνωρίζω επίσης και τις ε, δυσκολίες που περνάει η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή οικονομία. Επομένως ε, το ερώτημα είναι θεωρείτε γιατί για εσάς που εκπροσωπείτε αυτές τις βιομηχανίες θα πρέπει να είναι μια κόκκινη γραμμή. Δεύτερη ερώτηση. Πέρα από τη διαπραγμάτευση για την TTIP, υπάρχει συμφωνία με τον Καναδά. Εδώ δεν υπάρχει ο κίνδυνος εξαιτία της συμφωνίας με τον Καναδά να, μπορούμε, να, να μην μπορούμε να ασκήσουμε την ίδια πίεση στις Ηνωμένε Πολιτείες. Γιατί οποιοδήποτε consortium συμπεριλαμβάνει μια καναδική εταιρεία θα μπορούσε να ε, ε, υποφεληθεί από τις προβλέψεις της TTIP. Επομένως θα ε, αποδυναμωθεί η διαπραγματευτική μας θέση με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, μήπως μας πούνε ότι δεν θα ήθελαν να ε, μπουν καν στη διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, την τύπη για αυτά τα θέματα. Επίσης, η ευρωπαϊκή ναυπηγική μειοβιχανία πολύ υψηλής ποιότητας ε, πλοία και τεχνολογία. Μέχρι το 60%, μάλλον με τον περιορισμό του 60%. Το ερώτημα είναι το εξή, δεν θα μπορούσαμε εμείς να παρέχουμε υπηρεσίες σεβόμενοι το όριο του 60% που θέτουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και χρησιμοποιώντας εργαζόμενους από τις Ηνωμένε Πολιτείε τοπικά. Νομίζω ότι ίσω κάποιε από αυτέ τι ερωτήσει είναι καλύτερα να τι απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω εκείνε που αφορούν στη διαπραγματευτική μα τακτική. Σα Τόλτον. ευχαριστώ για τι παρουσιάσεις, ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Μα δείχνουν πόσο προστατευτικοί είναι, είναι, προστατευτικές είναι οι Ηνωμένες για την αγορά τους. Πρώτα απ' όλα, πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αλλάξουν την πολιτική του. Σίγουρα δεν θα τους πείσουμε να καταργήσουν την νομοθεσία, ούτε την Jones Act, ούτε τον Buy America. Αλλά πόσο ρεαλιστικό πιστεύετε ότι θα, μπορούσατε να τους, θα μπορούσαμε να τους πείσουμε να την τροποποιήσουν. Επίση, νομίζω ότι και από τις δύο παρουσιάσει μπορούμε να συναγάγουμε πόσο αυτού του τύπου οι περιορισμοί ε, πλήττουν τις επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο. Και γι' αυτό εκπλήσωμε από την, παρουσίαση του, από την παρέμβαση του τρίτου μιλητή από τα συνδικάτα που έλεγε ότι θα ήθελε να δει κάτι παρόμοιο στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες ε, ε, θέσει εργασία στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι αντιθέτω η άρση αυτών των περιορισμών θα δημιουργούσε θέσει εργασία στην Ευρώπη. Και έρχομαι στο θέμα που τίθεται, για την προστασία του καταναλωτή. Το σκάνδαλο τη Volkswagen από τι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε, όχι από την Ευρώπη γιατί γνωρίζουμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε όταν υπάρχει ένα πρόβλημα προστασίας του καταναλωτή ή προστασίας του περιβάλλοντος προτιμούν τη δικαστική οδό παρά την υιοθέτηση νομοθεσίας όπως συνήθως κάνουμε εδώ. Το ερώτημά μου είναι, είμαστε προκατελημένοι μήπως στην Ευρώπη και θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο να παραβιάσει κανείς την εργατική ή την παρεβαλλοντική νομοθεσία στις ΗΠΑ ή όντως ισχύει αυτό. Η ε, κυρία Κέπχαρτ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διοργάνωση της σημερινή ακρόαση γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα το οποίο πραγματεύεται και θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις και όχι τόσο ερωτήσεις. Η πρώτη, μεταξύ άλλων και για τα θέματα τα οποία ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Καταρχά λοιπόν, το 60% σχετικός περιορισμός σε ό,τι αφορά το Buy American Act σε ομοσπονδιακό επίπεδο ισχύει αυτό το ποσοστό. Και εξ όσων γνωρίζω υπάρχει και επιπρόσθετος περιορισμός σε επίπεδο πολιτιών. Αυτό ασφαλώς αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο, το, η συμφωνία που θα διαπραγματευτούμε θα είναι με το, με, τα, με το Ομοσπονδιακό κράτος, όχι με τις πολιτείες. Πώς λοιπόν θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να ανοίξουμε εμείς ε, τις δικές μας αγορές και μάλιστα σε εκεί να ανοίξει η αγορά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όχι όμως σε επίπεδο πολιτιών. Αυτό θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει σίγουρα να τεθεί. Ότι, δηλαδή, πόσο μεγάλη είναι η αρμοδιότητα και η ευθύνη των ε, πολιτιών και τι μπορούμε να κάνουν. Δεύτερη παρατηρήση. Εμεί στην πολιτική μα ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνεκτικοί. Να υπάρχει μεγάλη συνέπεια. Μα είπε η κυρία από τον ναυτιλιακό κλάδο ότι υπάρχει το, η εξή ένσταση. Στην αμερικανική αγορά έχουμε αμερικανικά μόνο προϊόντα. Και θυμάμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είχε γίνει μια τεράστια αμφιλεγόμενη συζήτηση για το θέμα του καποτάζ. Αν εμείς λοιπόν δεν είμαστε δεθμένοι να ανοίξουμε τον κλάδο αυτό, πώς μπορούμε να το απαιτήσουμε από τις ΗΠΑ και μήπως αυτό θα σήμαινε συνεκδοχικά ότι και εμείς θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή να θέσουμε υπό αμφισβήτηση και τις δικέ μα ρυθμίσει και μάλιστα τι ρυθμίσεις μεταξύ άλλων και για την προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιε είναι οι συνέπειε και για τα δική μα αγορά. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία με απασχολεί και αν θα μπορούσε να το σχολιάσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτο τώρα σημείο. Αυτό που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες που προβλέπουν ε, πολύ σύγχρονα κριτήρια για την ανάθεση τέτοιων συμβάσεων σε ό,τι αφορά την κοινωνική, οικολογική πτυχή και άλλα κριτήρια και σε ό,τι αφορά γενικότερα την προστασία των κοινοφιλών υπηρεσιών. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως προκειμένου να μην υπονομευθούν όλα αυτά από μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και με οποιονδήποτε άλλο εταίρο. Αυτό άλλωστε το έχουμε εκφράσει και σε διάφορα ψηφίσματα. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριο Κασπάρη. Αγαπητοί συνάδελφοι. Να συνεχίσω από αυτά που είπε στο τέλος η κυρία Γκέπχαρτ. Γιατί μεγάλο τμήμα του κόσμου ανησυχεί σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και σε ό,τι αφορά την Σύμβαση Εμπορικών Συμφωνιών ότι θα μπορούσε να προκύψει η δυτικοποίηση Στη ε, Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, υπάρχει ανησυχία για την δυτικοποίηση του τομέα υδροδότηση και στη δική μου πατρίδα υπάρχουν τέτοιε ανησυχίε. Αλλά θεωρώ ότι το σημείο εκκίνηση είναι ότι εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι συμφωνούν. Ούτε ένα συνάδελφο δεν έχω ακούσει που να είπε ότι θα συμφωνούσε με ένα TTIP που θα προέβλεπε ιδιωτικοποίηση κοινοφελών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η υδροδότηση σε ε, επίπεδο δημοτικό. Θα ήθελα να το μεταφέρουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα προς τα έξω, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανείς τίτη που να υπονομεύσει αυτού τους κλάδους. Μία συγκεκριμένη ερώτηση να κάνω όμως. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο κάποιος από τους πάνελίστες έχει αριθμητικά στοιχεία για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι αγορές δημόσιων προμηθειών. Γιατί όγκο μιλάμε, δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή συμμετοχή στη ΣΥΠΑ. Μάλλον, σε πόσο μεγάλος είναι ο κλάδος αυτός στη ΣΥΠΑ, πόσο μεγάλος είναι ο κλάδος αυτός στην Ευρώπη και ποια είναι η σχέση συγκριτικά μεταξύ των δύο κλάδων αυτών για να δούμε τι θα σήμερα αυτό ενδεχομένως και για ε, την αγορά εργασία μα. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Φόρντ. Αυτό το ερώτημα ενδεχομένω να μπορούσε να απευθυνθεί και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλοι δύο ομιλητέ. Η κυρία Γιακονσάρη είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Λίσα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε για το χρονοδιάγραμμα φαίνεται ότι, ότι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει μεγάλη αντίσταση σε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Το ίδιο είδαμε και με τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τις χώρες του Ειρηνικού. Και γνωρίζουμε ότι έρχονται και οι προεδρικές εκλογές. Και ε, από ό,τι έχει φανεί στην προεκλογική εκστρατεία, κανένας από τους υποψηφίους που ηγούνται το δημοσκοπήσεων ε, δεν είναι υπέρ αυτών των ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Οι περισσότεροι ε, καταφέρονται εναντίον τέτοιων συμφωνιών. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες αυτών των συμφωνιών, αλλά έχουν μια γενική εικόνα. Και αναρωτιέμαι μήπως θα ήταν καλύτερα να θέσουμε επιτάπητο στο θέμα των φορολογικών παραδείσων. Το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως σημαντικότερο από τις σιδηροδρόμους ή άλλα πράγματα από αυτά που ακούσαμε. Ο κύριος Βίνκλερ, ο οποίος είναι ο τελευταίο ομιλητή, γιατί θα ήθελα και οι εμπειρογνώμονε μετά να πάρουν το λόγο και να έχουν ε, ε, αρκετό χρόνο. Και επίση να διευκρινίσω ότι κάποιε από τι ερωτήσει που θέτατε, τη συνάδελφοι, μάλλον είναι προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης σήμερα. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Εδώ υπάρχουν διαφορές στα κριτήρια και στις ε, νομοθεσίες, αλλά οι δημόσιες συμβάσεις και οι δημόσιες προμήθειες είναι ξεκάθαρα ένα πολιτικό θέμα και σωστά αναφέρατε ότι αναμένουμε και επίσκεψη του Πρόεδρου Ομπάμα στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή τον Ιανουάριο του 2017 γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα θα παραδώσει στον επόμενο Πρόεδρο. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που σχετίζεται με τις δημόσιες προμήθειες, όχι μόνο, αλλά και με αυτέ, και είναι οι απαιτήσει όσον αφορά τι θεωρήσεις, η βίζα. Ε, και εγώ θα ήθελα λοιπόν να ε, θέσω το θέμα ως εξής, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες συνεχίζεται να ζητείται από τους πολίτες τους να ε, έχουν θεώρηση όταν ε, επισκέπτονται τις ΗΠΑ για να μεταβούν στις ΗΠΑ και αυτό επηρεάζει και τους σιδηροδρόμους και την ε, ναυπηγική βιομηχανία. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν από τους προσώπους αυτών των δύο βιομηχανιών να μας πούνε αν και πώς επηρεάζονται. Και δεν αφορά μόνο τη Ρουμανία, αλλά και άλλες χώρες αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα επίσης να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό και επίσης για το εάν θα τεθεί το θέμα αυτό στον πρόεδρο Ομπάμα όταν επισκεφτεί την Ευρώπη σε λίγες ημέρες. Έχω και εγώ μια ερώτηση για την κυρία Σέν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάσαμε πρόσφατα ένα νέο ε, πλοίο για έρευνα στην Αρκτική θάλασσα. Εάν ένας επιστήμονας από τις Ηνωμένε Πολιτείε. ήθελε να αγοράσει ένα παρόμοιο πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα τους το επιτρέπεται αυτό δηλαδή ένα πλοίο το οποίο θα είχε κατασκευαστεί με την ίδια τεχνολογία, με το ίδιο σχέδιο σε ένα ναυπηγείο στις, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο για να χρησιμοποιηθεί για έρευνα στον αρκτικό κύκλο. Αυτό θα επιτρεπόταν ή θα απαγορευόταν βάσει την Αμερικανική νομοθεσία. Θα δώσω το λόγο με την αντίστροφη σειρά από αυτήν με την οποία μιλήσατε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις όλοι. Ο κύριος Μπασό λοιπόν ξεκινούμε. Εν συντομία. γιατί τα συνδικάτα των ΕΠΑ είναι τόσο προστατευτικά. Γιατί είχαν πάρα πολύ κακές εμπειρίες με προηγούμενε ε, συμφωνίε ελευθερού εμπορίου στην, ε, στις Είχαν πολύ κακέ εμπειρίες με την ΑΦΤΑ, με την οποία ήταν αντίθετη. Είναι αντίθετη τώρα ως προ το TTIP. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να προστατεύσουν την αγορά τους. Για μας δε το θέμα της αμοιβαιότητας είναι πολύ βασικό. Αν οι ΙΠΑ δεν ανοίξουν την αγορά των δημοσίων προμηθειών τους, γιατί δεν θα ανοίξουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα. Και θα δούμε κατά πόσο θα είναι πρόθυμοι οι Αμερικανοί να το συζητήσουν αυτό εξ όσων γνωρίζω, στις άλλες συμφωνίες ελευθερεμπορίου προστατεύσαν πολύ την αγορά δημοσίων προμηθειών. Αλλά εμεί, ε, ως σημείο φετηρία έχουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε πετύχει καλά πρότυπα, κοινωνικά πρότυπα και ούτω καθεξής στι ε, δημόσιες προμήθειές μας και δεν θέλαμε αυτό να υπομονωμευτεί σε καμία περίπτωση από συμφωνίε ελευθερού εμπορίου. Η κυρία ευχαριστώ. Εγώ τρεις ερωτήσεις ε, ε, έχω να απαντήσω, θεωρώ. Καταρχάς, το θέμα του βυθακόρου. Νομίζω ότι στην αρχή της παρουσίασής μου διευκρίνησα ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση γιατί εμείς είμαστε ναυπηγοί. Δεν είμαστε ούτε κάτοχοι, ούτε ιδιοκτήτες, ούτε ε, εταιρεία διαχείρισης ε, σκαφών. Ρωτήσατε λοιπόν τι γίνεται με τις ε, υπηρεσίε μυθοκόρηση. Δεν μας αφορά αυτό, εμείς κατασκευάζουμε μόνο. Η βυθοκόρη και άλλα τέτοια σκάφη είναι μια λυπηρή ιστορία. Γιατί τρεις φορές έχουν τιμωρηθεί στην, ε, στη ΣΥΠΑ. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό δεν μπορούν να απολύσουν πάνω από το 40%. Σε ό,τι αφορά το Jones Act, πάλι υπάρχει ε, σχετική προστασία και στις ΗΠΑ πάντα είναι η διακτησία της κυβέρνησης. Άρα πάντα διακατέχονται και ε, ελέγχονται, μάλλον υπόκεινται στις προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Δεν βλέπω λοιπόν καμία προοπτική να αλλάξει τον ο νόμος. Ύστερα, μου ζητήσατε να υπολογίσουμε τον όγκο τη αγοράς δημοσίων προμηθειών. Εύκολο αυτό. Γιατί στην παρούσα φάση είμαστε σε μηδενικό ποσοστό. Γιατί οι ΙΠΑ δεν έχουν τεχνολογία, δεν έχουν σκάφη. και δεν μπορούν να καλύψουν καν τι δικέ του ανάγκε. Πόσο μάλλον τι ευρωπαϊκέ. Εμεί δεν έχουμε πρόσβαση στη δική του αγορά. Άρα, μηδέν είστε πελικό. Τώρα για το παγοδραστικό που ρωτήσατε. Φυσικά παρακολουθούμε στις ειδήσει το τι μπορούσε, θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην, στην Γερμανία, στην ε, Γαλλία, στη Φιλανδία. Υπάρχει τεχνογνωσία για την αφήγηση υποδραστικών και ασκούμε λόμπι και στην ακτοφυλακή στις ΙΠΑ για να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους πούμε ότι κοιτάξτε στην Ευρώπη έχουμε τεχνογνωσία και αν έχετε και προβλήματα χρηματοδότησης μπορούμε πάλι να βοηθήσουμε αλλά η αμερικανική ακτοφυλακή και το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει εξαίρεση για την ακτοφυλακή αν υπογραφεί από τον Πρόεδρο, αλλά θα πρέπει να αποδεχτεί η κατεπίγουσα Α, Υπάρχει μια μικρή δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να πιστούν. Και αυτό υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητα από το TTIP. Ελπίζουμε λοιπόν να μην συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε από αυτή τη μικρή εξαίρεση για τις πωλήσει στον κλάδο αυτό. Ευχαριστώ ο κύριος Ευχαριστώ. Τα μέλη της UNIFE δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ευτυχής γι' αυτό, αλλά βέβαια δεν μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δημόσιες προμήθειες κάθε φορά που υπάρχει προκήρυξη. Η πρότασή μας λοιπόν προς την Επιτροπή Ομάδα Διαπραγμάτευσης είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο θα πρέπει να μην δεχθούμε το local hiring που λένε οι Αμερικανοί, δηλαδή τις προσλήψεις ε, ντόπιων εργαζομένων. Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση του Καναδά θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από αυτή γιατί δεν μιλούσαμε για local contact αλλά για local values αυτές και ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Και... Ο πρόεδρος. Η πρόεδρος. Τη σκητάλη τρώει το δεύτερο πάνελ, ο κύριος ε, Λάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε για σωρό προβλήματα, αλλά και ε, περιορισμούς, το John Jack και άλλα νομοθετήματα, ακόμα και προβλήματα που ξεκινούν από εδώ, από την Ευρώπη, όσον αφορά το τι θα γίνει με τις δημόσιες συμβάσεις, τι θα γίνει με τις απαιτήσει σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. Τώρα έχουμε το, ε, τη δεύτερη ομάδα ομιλητών, δεύτερο πάνελ και θα πρέπει να δούμε το πώς θα εξασφαλίσουμε το να υπάρχει διαφάνεια, το να μην υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις για τις ε, ε συμβάσεις προμηθειών και επίσης το πώς θα τηρούνται και οι προϋποθέσεις της κοινωνικής πολιτικής. Έχουμε και εδώ προσκεκλημένους ε, ειδικού βεβαίως είναι βασικά νομική, γιατί είναι νομικό το θέμα το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις εγγυήσεις αποκλεισμού ε, του, των ζημινών ε, διακρίσεων και των κοινωνικών ε, προτύπων. Ξεκινώ με την ε, δόκτωρα Καμάλα Νταβάρ που είναι λέκτορ σε θέματα διεθνούς εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Σάσετ. Έχετε το λόγο ευχαριστώ που με καλείστε εδώ και βλέπω ότι κυρίως ε, μιλάτε όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και όσον αφορά τις ε, συμβάσεις. Εγώ όμως τώρα θέλω να στιάσω την προσοχή μας στο τι γίνεται με αυτές τις εμπορικές συμφωνίες γιατί εκτός από την εμπορική πτυχή έχουμε και το θέμα της διακυβέρνησης και ίσως ε, α, εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να αποσπάσουμε κάποια αποτελέσματα χωρίς τα προβλήματα της πρόσβασης στην αγορά. Οπότε θα σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Και έχουμε εδώ πέρα κάποια, κάποιες αρχές, ε, ακριβώς όπως και στο εμπόριο και πρέπει να δούμε το πώς αυτές οι αρχές για την διακυβέρνηση είναι δυνατόν να μας οδηγήσει ε, σε κάποιο είδους ε, ωφέλεια για το ευρύτερο κοινό. Και οπότε θα πρέπει να δούμε για ε, ε, το πώς θα άρουμε κάποιους de facto φραγμούς ή στο, ε, στο εμπόριο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όπως προανέφερα εδώ έχουμε δύο πτυχές. Την εμπορική πτυχή, de jure, ε, σε σχέση με την πρόσβαση σε σχέση με την ισότητα μεταχείρισης και επίσης τις ε, διαπραγματεύσεις ε, που καθορίζουν τη συνέχεια. Αλλά υπάρχει και η πτυχή της διακυβέρνησης που είναι φραγμός de facto και όχι de jure. Οπότε έχουμε, θα πρέπει να έχουμε ε, διαφάνεια, θα πρέπει να έχουμε υποχρέωση λογοδοσίας και πάρα πολύ σημαντικό είναι το τι γίνεται με τη σύγκρουση συμφερόντων και την διαφάνεια. Ε, οπότε οι διαπραγματεύσει μας οδηγούν στη ρύθμιση του πόσο ρυθμίζεται η προσβασιμότητα στην αγορά. Οι βασικές πτυχέ είναι αυτές, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ε, δεσμενεί διακρίσει για τους προμηθευτές, θα πρέπει να ε, έχουμε ε, αυτή την, ε, την αποφυγή διάκρισης για αγαθά και υπηρεσίες, να υπάρχει διαφάνεια στο σύστημα και επίσης να υπάρχει διαδικαστική ε, δικαιοσύνη για τους εν δυνάμει και τους εν ενεργεία προμηθευτές. Βλέπουμε ότι δεν είναι διαφθορά η διακριτική μεταχείριση, αλλά θα πρέπει πάλι να δούμε τι γίνεται με το πώς θα αποκλείσουμε ε, το να υπάρχει αυτό το ψεγάδι τη δυσμενής διάκριση. Τώρα για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την εύνοια ε, της εσωτερικής αγοράς των προμηθευτών από την ίδια χώρα. Θα πρέπει επομένω να δούμε ότι το 1999 υπήρχαν στοιχεία που ανέδειξαν το ότι πριν την οδηγία όλες οι συμβάσεις των τοπικών αρχών πήγαιναν σε ντόπιου. Οπότε βλέπουμε ότι ευνοούνται οι ντόπιοι. Οπότε είναι σημαντική αυτή η οδηγία γιατί έρει αυτούς τους ε, φραγμούς όσον αφορά την αγορά των προμηθειών στην Αμερική. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ομοσπονδιακός νόμος, αλλά συνήθως γίνονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι προμήθειες υπάρχουν διάφοροι φραγμοί στο εμπόριο που είναι de facto. Τώρα η εύνοια του ντόπιου το εννοεί, αλλά έχουμε και τους φραγμούς de jure που δεν τους κοιτάζουμε τώρα. Αυτό που θέλω τώρα να δούμε είναι ότι αυτή η εύνοια δεν οφείλεται σε ε, νομοθέτημα ή σε τιμολογική πολιτική αλλά στο ότι η ντόπιοι πολιτικοί ενδιαφέρονται να ευνοήσουν τους ντόπιου. Άρα ε, μεγάλο πρόβλημα είναι το να μην υπάρχει διαφάνεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για τις ΜΜΕ, γιατί δεν έχουν τους πόρους για να μπορέσουν να καλύψουν ε, τα, τα απαιτούμενα. Αλλά ε, έχω εδώ ένα συνάδελφο που θα σας το αναλύσει αυτό. Άρα μιλούμε για διαφάνεια σε όλη την διαδικασία της προμήθειας, αλλά και στους κανόνες των διαγωνισμών. Ποιος κέρδισε το διαγωνισμό, γιατί κέρδισε και δεν έχουμε αρκετά στοιχεία όσον αφορά την αγορά των προμηθειών, αλλά είναι φραγμός όταν απουσιάζει η διαφάνεια. Να δούμε τώρα τι γίνεται με την ε, διαφάνεια εδώ. Το θέμα είναι η προβλεψιμότητα. Είναι η ηλεκτρονική διαγωνισμή. Να, κοιτάξτε τι γίνεται στην ε, Σλοβακία. Το 2009 είχαν κάποιες, κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις για περισσότερη διαφάνεια. Οπότε από 2,3 πήγε στο 3,6 όσον αφορά τις προσφορές. Με αυτό ε, σημαίνει περισσότερο ανταγωνισμό, σαν τα χρήματα τόπο, καλύτερες τιμές, περισσότερη καινοτομία αλλά και επιλογή. Τώρα για να δούμε άλλους φραγμούς de facto. Είναι η διαφθορά. 20% ε, είναι, εκτιμάται ότι είναι οι διαρροές από αυτόν τον λόγο γιατί έχουμε εκ των προτέρων έλεγχο για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κλπ. Υπάρχει όμως και μηχανισμός ε, εξόδικού συμβιβασμού εκ των υστέρων και προχωρούμε με ε, κάποιες ε, εξελίξεις σε επίπεδο ΠΟΕ, Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, επί τη βάση του συστήματος της Νοτιού Κορέας. Εκεί υπάρχει ηλεκτρονικός διαγωνισμός, σύστημα e-procurement και μιλάμε για τον κρατικό τομέα ότι το κόστος εδώ είναι 1,4 δις και ο ιδιωτικό 6,6 δις. Ναι, και ε, αφού δούμε τι δρόμο θα πάρει το TTIP. Άρα, ε, να δούμε ποιες είναι οι θετικές ρυθμιστικές συνέργειες. Έλεγχο της ακυριότητας, της μη διακριτής μεταχείρισης, έλεγχο της διαφθοράς. Και έτσι μπορούμε τα δημόσια αγαθά να τα καλύψουμε, αυτό θα είναι για τον κόσμο. Ε, πάρα πολύ καλό. Μιλάμε για τους δημόσιου πόρους για όλους. Δεν μπορούμε αυτά να τα εξαντλήσουμε, μπορούμε να τα ε, μοιράσουμε. Και εν συμπεράσματι, όλοι γνωρίζουμε ότι στο TTIP θα πρέπει να καλυφθεί η σωστή διακυβέρνηση με το σύστημα εγγεμένου προτιμήσεων συν και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα διάφορα με τους διάφορους φραγμούς de facto και de jure ε, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε ΠΟΕ και τι γίνεται στην Συμφωνία ΣΕΤΑ. Είναι θέμα που θίγει ανταγωνισμό, ε, για την ανάπτυξη, για τις τιμές. Οπότε θα βάλουμε τελεία λέγοντας ότι τα θέματα διακυβέρνησης έχουν δυναμητιστεί από το πρόβλημα και τη μεγάλη προστασία στον χρόνο την προβασιμότητα στην αγορά. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Ναι, καλύπτουμε όλες τις χώρες του κόσμου και όχι μόνο κάποια συγκεκριμένη ε, χώρα που έχει προθωμένη βιομηχανία έχουμε προβλήματα ακόμα και εδώ βλέπετε από πλευράς τεχνολογίας και πληροφορικής γιατί δεν λειτουργεί η οθόνη που είναι πίσω μου οπότε έχουμε μόνο τη μία οθόνη απέναντί μου συμπαθάτε με αλλά τι να κάνουμε ωραία τώρα αυτό ήταν η άποψη από πλευράς των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων ε, στην Ευρώπη και τώρα έχουμε όμως ε, και κάποιον Αμερικανό εμπειρογνώμονα και ανυπομονώ να ακούσω το εάν συμφωνεί. Είναι ο καθηγητής ε, Γιάκινς από το Πανεπιστήμιο George Washington. Ε, στην νομική σχολή εργάζομαι και είμαι συνδιευθυντής όσον αφορά το πρόγραμμα του δικαίου των συμβάσεων. Ε, σε επίπεδο ΙΠΑ είμαστε πρωτοπόροι και με μεγάλη μου χαρά ε, ήρθα εδώ να σας τα πω. Next slide, negotiations... Οι διαπραγματεύσεις για το TTIP μεταξύ Ένωσης και ΕΠΑ έχουν σημαδευτεί από σημαντικές διαφωνίες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά των προμηθειών. Μία προσέγγιση θα ήταν να ζητήσουμε το να υπάρξουν κάποιο είδους ενισχύσεις ομοσπονδιακές. Και αυτό θα ήταν μια ε, πολιτική κατά της ε, δυσμενούς διάκρισης και μιλάμε για 600 δις. Ε, την κρατική ενίσχυση, τη λέμε, αυτά τα 600 δις, τα, λέμε εμείς ενισχύσεις στις ε, κρατικές επιδοτήσεις που λέτε εδώ στην Ευρώπη. Και τώρα για αυτά τα 600 δις είπαμε ότι οι δικαιούχη απαγορεύεται να δείχνουν κάποια γεωγραφική προτίμηση. Και εάν αλλάξει κανείς μόνο τρεις λέξεις σε αυτό τον νόμο, δηλαδή το ε, πολιτεία ή ντόπιο. Και βλέπουμε ότι όταν κάποιος δικαιούται αυτή την ενίσχυση δεν θα πρέπει να, ε, να προβαίνει σε αυτή τη διάκριση και άρα ανοίγει την πόρτα για τα της Πρόκειται για νομοθεσία προέρχεται από τον Λευκό Οίκο, δεν υπάρχει καμία, κανένας ε, περιορισμός όπως το Τζον Ζακ. Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν να ενθαρρύνουμε την ρυθμιστική συνεργασία και έτσι να ελιάνουμε τις διαφορές μας για την ασφάλεια, την βιωσιμότητα, αυτά που θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτό θεωρώ ότι είναι εφικτό. Η εναρμόνιση αυτή ε, περιέχεται και στην πρόταση της Επιτροπής για τον συντονισμό στα ρυθμιστικά. Και έτσι θα ελεγχθούν διαφορές μεταξύ ΙΠΑ και Ένωσης. Τώρα δε έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή πρόταση στα πλαίσια του TTIP. Είναι μια ευρεία πρόταση. Διατυπώθηκε πριν από ένα μήνα και πρόκειται για συνεργασία σε όποιον τομέα θεωρείται κοινού ενδιαφέροντος από τις ρυθμιστικές αρχές. Οπότε, αυτή η πρόταση μπορεί να μας οδηγήσει σε συνεργασία στις προμήθειες. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να ένα παράδειγμα. Από το Υπουργείο Αμήνης. Είναι ένας κανονισμός και αναφέρεται σε μη διαβαθμισμένες πληροφορίες όσον αφορά τη συνεργασία με κάποιους προμηθευτές. Εδώ προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ένα πρόβλημα ασφάλειας. Εδώ έχετε το ISO για τα πρότυπα και εμείς έχουμε αυτά τα πρότυπα που βλέπετε εδώ από το Εθνικό Ίδρυμα ε, Προτύπων και Τεχνολογίας και αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ένας ξένος Ευρωπαίος ε, προμηθευτής να προτείνει μια λύση κυβερνοασφάλειας όχι βάσει του ISO αλλά βάσει των δικών μας προτύπων. Βάσει της υπηρεσίας συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας. Να ένα ε, παράδειγμα του που μπορείτε να χτυπήσετε, που μπορείτε να προτείνετε. Και έτσι Μπορεί κάποιος Ευρωπαίος να προτείνει κάποια λύση για αυτά τα προϊόντα που είπαμε και έτσι σας ξανήγεται η αγορά της κυβερνοασφάλειας. Πάντως έχουμε και άλλους κανονισμούς για κυβερνοασφάλεια που δεν είναι όπως ο κανονισμός αυτός. Δεν δηλαδή τέτοια, δεν ξανοίγονται σε τέτοιες λύσεις προς τους ξένους τώρα. Άλλο παράδειγμα που έχει σχέση με την αρμόνιση και εδώ μπορεί να έχουμε ένα αρμόνιση μας μεταξύ των μεν και των δε είναι αυτού του είδους η, η βιωσιμότητα που οδηγεί σε ολοκλήρωση integrating sustainability και εδώ προβλέπεται από δικό μας και από δικό σας ε, νομοθέτημα η οικολογική ετικέτα. Υπάρχει διαφορά βέβαια στην ετικέτα σε κάθε πλευρά, αλλά με αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με την απόφαση Μαξ Χάβρα, ρυθμίζεται το πρόβλημα αυτό. Η απόφαση αυτή Max Χάβρα λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές οικολογικές ετικέτες άπαξ και κάποιο εξηγήσει το θεμέλιο αυτών. Οπότε μπορεί να ε, χρησιμοποιεί διαφορετική ετικέτα, αν κανείς το εξηγεί. Οπότε θα μπορούσε αυτό να περάσει εάν περιληφθεί στη συμφωνία TTIP. Σωστή προσέγγιση και αυτό τώρα αποτελεί δίκαιο, αποτελεί νομολογία. Παρά τις διαφορετικές ετικέτες, επομένως έτσι ξανοίγεται πάλι προσβασιμότητα να, ένα παράδειγμα. Η απόφαση Max Χάβλα. Πώς μπορούμε να έχουμε συνεργασία και εναρμόνιση. Και εδώ βάζω τελείω και σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Εκείνοι που θα αφηληθούν θα έπρεπε να αφηληθούν από την εξάλληψη των δυσμενών διακρίσεων στις δημόσιες συμβάσεις θα, θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πάνελ μας ε, σήμερα, κυρία Σίτσκε Τικχούτ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούσαμε για το πώς μπορεί να γίνει περισσότερο διαφανή η διαδικασία των δημοσίων προμηθειών και πώς αυτό ευνοεί και τα δύο μέρη. Αυτό γίνεται όταν δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της διαδικασίας της κυβέρνηση και όχι τόσο στην πρόσβαση στην ώρα. Εγώ θα στεθώ στο πώς μπορούν να αφαιρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ένα τέταρτο των ε, επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η Ένωσή μας εξάγουν. Ε, πρώτης προορισμός είναι η Ευρώπη και δεύτερος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένω, ε, ε, με τη βελτίωση της νομοθεσίας θα μας δοθεί η δυνατότητα να αυξηθεί και ο όγκος των εξαγωγών αλλά και να γίνουν αυτές προς περισσότερες χώρες. Η στόχη είναι όσον αφορά τη διαφάνεια η εξή. Πρώτα απ' όλα μια διαφάνεια ως προς τις ε, ευκαιρίες που υπάρχουν, δηλαδή ε, να, να είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς ότι έχει υπάρξει μια προκήρυξη. Ε, ανεξαρτήτως ε, της αξίας τους σύμβασης, γιατί κάποιες συμβάσεις μικρότερης αξίας είναι εκείνες που ενδιαφέρουν περισσότερο τις μικρομεσαίες εταιρείες. Σύμφωνα με, εμά, τη συμφωνία TTIP προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα πόρταλ, μια πύλη πληροφοριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό θα αυτή του τύπου διαφάνεια θα μπορούσε να γίνει μέσω αυτού. Επίσης χρειαζόμαστε ξεκάθαρα κριτήρια για την επιλογή, για τη βαθμολόγηση των προσφορών. Να γνωρίζουν ποιο κέρδισε τελικά, σε ποιον κατακυρώθηκε η σύμβαση και γιατί. Και κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι η δυνατότητα και η περίοδος κατά την οποία μπορεί κάποιος να υποβάλει ένσταση. Ορισμένες ε, αναθέτουσες αρχές μερικές φορές το αποφεύγουν αυτό, καταφέρνουν να μην δώσουν τη δυνατότητα στους προσφέροντες να υποβάλουν ενστάσεις όταν το θέλουν. Θα σας δώσω το παράδειγμα ενός συστήματος που ε, λειτουργεί, η B-Cloud και το οποίο μας τη δυνατό, έχει δώσει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται ισότιμα, μεγαλύτερες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να προσαρμόζονται γρήγορα, κάτι που βοηθάει όταν υπάρχει διαφάνεια ε, στην ανάπτυξη στο να λειτουργούν αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν ε, εταιρείε μικρές ε, στην Ιρλανδία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής και έχουν καταφέρει να πάρουν συμβάσεις στις ΗΠΑ για τα πληροφορικά συστήματα των ε, φυλακών. Υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας με μεγαλύτερες εταιρείες, αλλά αυτό δεν είναι πάντα η καλύτερη ε, επιλογή. Όταν κανείς μπορεί να είναι πιο αυτόνομος, ε, έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί ευθέως και μεγαλύτερες εταιρείες σε όλα τα μέρη της TTIP θα έπρεπε να προωθήσουμε τη διαφάνεια και στο κεφάλαιο που αφορά στις ε, συμφωνίες, στο ελεύθερο εμπόριο και στο κεφάλαιο που αφορά στις μικρομεσαίες. Τέλος, οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα μέρος της Διατλαντικής Συμφωνίας, της συμφωνίε εμπορίου με τι Ηνωμένε Πολιτείε και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει μπορούν να επωφεληθούν συνολικά από την αγορά. Ε, Αντιθέτω, εάν η TTIP δεν ε, δώσει τη δυνατότητα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει να ε, δραστηριοποιηθούν στι δημόσιε συμβάσει, θα μπορούσε αυτό να είναι πολύ κακό για τι ίδιε. Θέλουμε λοιπόν η TTIP να οδηγήσει σε ένα άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων. Μιλώντας τώρα για το ζητήματα της διακυβέρνηση και πάλι η διαφάνεια είναι το πιο σημαντικό, βοηθάει και την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα κάνουμε το γύρο των ερωταπαντήσεων. Έχουμε 20 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας. Ε, οι ερωτήσεις λοιπόν να διαρκέσουν ε, μέχρι ένα λεπτό. Ο κατάλογος των ομιλητών, παρακαλώ. Έξι ομιλητές. Έξι άτομα έχω ζητήσει το λόγο. Ο πρώτος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητές που προωθούν τα θέματα διαφάνειας, γιατί συμφωνώ και μου άρεσαν και τα παραδείγματα της τελευταίας ομιλητρίας, η οποία ε, μίλησε για θέματα στη Σλοβακία. Να σας πω ότι εγκρίναμε το σχετικό νομοσχέδιο, ότι οι δημόσιες συμβάσεις και σχετικές ε, συμφωνίες ισχύουν μόνο αν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Μόνο με αυτό λοιπόν μειώσαμε κατά 14% τις δαπάνες Στι δημόσιε συμβάσει σε ένα μόνο έτο. Τον κύριο Γιούκενς λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω ο οποίο ενδεχομένω θα ξέρει πολύ καλύτερα από την εμπειρία του, κατά πόσο ε, πιστεύετε ότι τέτοιου είδου ρήτρε θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και να μπουν στην ε, Αμερικανική νομοθεσία για να αυξήσουν τη διαφάνεια ή ενδεχομένω να μπουν και στην Συμφωνία TTIP. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους, αλλά θα ήθελα να κάνω και μια γέφυρα μεταξύ των δύο πάνελ. Γιατί πιστεύω ότι οι Ευρωπαϊκή δήμοι και οι τοπικές ε, αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να είναι σημαντικό ε, μέσο προκειμένου να δοθούν και τοπικά ε, κίνητρα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και για να θέσουν οικονομικά πρότυπα. Κοιτώντα λοιπόν το ζήτημα αυτό και τα θέματα που, έστελε, που έθεσε ο πρώτος ομιλητής, ανακύπτει το εξή ερώτημα. De facto, αυτό ισχύει. De jure όμως στις δημόσιες ε, προμήθειες υπάρχει κάποιος ε, κινητηρίος μοχλός για να βάλουμε τους ευρωπαϊκούς δήμους και κοινότητες στο επίκεντρο. Κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ, ήταν αρκετά ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό. Αλλά αν οι πολιτείε τη ΗΠΑ δεν καλύπτονται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, πώς ε, μπορεί να αλλάξει μια ανταγιούρε ρύθμισε την κατάσταση de facto. Ευχαριστώ πολύ. Η ΕΜΑ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και εγώ τους ομιλητές. Οι δημόσιες προμήθειες ε, έχουν ένα τεράστιο δυναμικό, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες μας. Πολλά έχουμε να κάνουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει Πολύ ευαίσθητη η σημερινή φάση. Αλλά με εντυπωσίασαν οι παρουσιάσεις όλων των ε, ομιλητών μας σήμερα. Να ρωτήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον έχει σκεφτεί αυτέ τι προτάσει που ακούσαμε από του πανελίστε σήμερα το πρωί και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτά που μα είπε ο πολύ γενναίο ε, εκπρόσωπο των ΗΠΑ για την πολιτική στην Αμερική. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε το θέμα της διαφάνειας, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι και για το που βρισκόμαστε κι εμείς. Μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι αυτή την εβδομάδα υποτίθεται ότι όλοι θα είχαμε εφαρμόσει τη σχετική οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά μόνο το ίμιση των κρατών μέλων το έχουν πράξει αυτό. Άρα θα πρέπει, εφόσον ζητάμε πιο πολύ διαφάνεια, να εξασφαλίσουμε ότι ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες για τη διαφάνεια και εμείς εδώ. Σε ό,τι αφορά την προβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εξέβρεση υποψηφίων, Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ε, κόμβος που να διατεθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα ήθελα να ακούσουμε και αυτά που έχει να μας πει ο συνάδελφος του FSP. Ευχαριστώ. Η Έμα. Ευχαριστώ και εγώ να συγχαρώ τους ομιλητές και έχω κάποιες ερωτήσεις για εκείνους. Για τον κύριο Γιάκινς. Πρωτή για τη πρώτη για οικονομία της αγοράς ελεύθερο το με το τότε πώ να τον έχετε προστατευτικού νόμου. Ποιο είναι ο λόγο ύπαρξη. Πώ πώς, πώς εγκρίθηκαν αυτοί οι νόμοι. Τα λόμπι είναι τόσο ισχυρά που εμποδίζουν τους πολιτικούς να λάβουν αποφάσεις που είναι σύντονες με το πνεύμα της χώρας. Τώρα κύριε Νταβάρ, πολύ καλά τα εξηγήσατε και συμφωνώ μαζί σας όμως νομίζω ότι θα πρέπει όσον αυτή διακυβέρνηση να δούμε τι θα γίνει και με την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων. Αυτό απουσιάζει. Δηλαδή να δούμε, κυρία Νταβάρ, τι είδους εταιρείε αναλαμβάνουν αυτά τα προγράμματα και τα έργα. Αφού θέλουμε να υπάρχει ε, κοινωνική ευθύνη, θα πρέπει επομένω ο κόσμος να ξέρει ότι αυτές οι επιχειρήσεις ε, ε, συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια. Τώρα, για την κυρία Ντεχρόντ, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, και στη δική μου χώρα όλες οι επιχειρήσεις ε, μπορούν να προσφύγουν στην ε, δικαιοσύνη σχετικά με τους ε, διαγωνισμούς υπάρχει δηλαδή δικαίωμα προσφυγής αλλά πάντως αυτό το δικαίωμα προσφυγής συνοδεύεται από κάποιες υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Θα πρέπει δηλαδή να είναι γνωστό το αν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Ο Γιώαχημ και εγώ έχω δύο ερωτήσεις γιατί ένα πράγμα δεν μου ταιριάζει με όλα όσα έχω ακούσει από τον οικονομικό κλάδο. Το κατά πόσον ε, οι δημόσιες προμήθειες πραγματικά ωφελούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί η δική μου εμπειρία στη Γερμανία σε ό,τι αφορά τις τοπικές ε, προμήθειες είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ε, ε κάποια δυνατότητα να συμμετέχουν και να παίρνουν τέτοιε σε συμβάσει. Όχι επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια, αλλά επειδή δεν είναι ανταγωνιστικέ σε σχέση με του μεγάλου ομίλου και είναι σε μερικτική θέση συχνά. Αν δεν ενισχυθούν τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Άρα υπάρχει κάποια στατιστική για το πώς ε, έχει αλλάξει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους ε, ε, των δημοσίων συμβάσεων, γιατί στην Ευρώπη έχουμε εδώ και καιρό ανοιχτές ε, αγορές δημοσίων προμηθειών. Και θα ήθελα να ξέρω τι ισχύει συγκεκριμένο. Ένα δεύτερο στοιχείο όπου θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε λίγο παραπάνω, θεωρώ, είναι το εξής. Οι ελεύθερες αγορές δημοσίων συμβάσεων δικαιολογούνται με το επιχείρημα της ε, μείωσης των εξόδων, των δαπανών. Αλλά υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα από πλευράς, ε, για παράδειγμα, οικονομικής, κοινωνικής, οικολογικής νομοθεσία. Δεν είναι μόνο το κόστος, λοιπόν, που παίζει σημασία, αλλά και το ποιε αξίε θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο των δημοσίων προμηθειών. Και θεωρώ ότι με τι δημόσιε προμήθειε έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να τα προωθήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. επόμενο. η κυρία Σανσαραβά. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητέ για την παρουσίασή τους. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό ως βάση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις μετέπειτα διαπραγματεύσει Αυτό το ενδιαφέρον που μας είπε η κυρία Νταχρότ και συμφωνώ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει θα πρέπει να είναι οι πρωταθλητέ του TTIP Γιατί κάποιε φορέ παρουσιάζεται ότι θα είναι μεγάλε επιχειρήσει, οι μεγάλοι όμιλοι αυτοί που θα ωφεληθούν. Αλλά πείτε μα κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Πώ έχει σήμερα η κατάσταση σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και σε ό,τι αφορά την ΕΠΑ. Αν υπάρχουν όντω ε, ε, επιτυχίε ε, στην αγορά δημοσίων προμηθειών και αν έχετε και αριθμητικά στοιχεία ενδεχομένω να μα παρουσιάσετε. Κυρία Φόρτ. Σύντομα. Θέλω να δούμε τι γίνεται με τις των αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε ε, να έχουμε τα ICT γιατί χρησιμοποιεί η Ευρώπη τα πρότυπα ISO και οι έχουν τα δικά του πρότυπα. Μήπω εμεί έτσι δημιουργούμε φραγμού όσον αφορά τη διαδικασία προτυποποίησης και έτσι δημιουργούμε προβλήματα για το μέλλον. Δεν ξέρω, μήπως ε, θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι ε, ε, προσκεκλημένοι μας να μας πούν πώς το βλέπουν αυτό για, τους, για, την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για να δούμε πώς μπορούμε να αναθεωρήσουμε τόσες σχήμες για την πρωτοβουλία εδώ στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος, κ. Νταβάρ, μας μίλησε για τον ΩΣΑ που είχε λέει 25% των προσφορών σε σχέση με την διαφάνεια, με συγγνώμη με την διαφθορά. Οπότε αυτό το πρόβλημα σοβεί και στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Θα ήθελα να μου μιλήσουν για αυτό το πρόβλημα επομένω και οι τρει ε, ομιλητέ μα. Και τώρα θα ακούσουμε τι ε, απαντήσει και ξεκινούμε με την αντίστροφη σειρά. Κυρία Δεχρόντ πρώτη. Ευχαριστώ. Εγώ έχω κρατήσει τρεις ερωτήσεις που απευθύνονταν σε μένα. Όσον αφορά πρώτα απ' όλα το κατά πόσον δημοσιοποιούνται οι δημόσιες συμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε ζητήσει να, να δημιουργηθεί αυτό το ε, πόρτερ πληροφόρησης και μέσω αυτού θα μπορούσαν να δημοσιοποιούνται και να είναι εύκολο να βρεθούν οι διάφορες προκηρύξεις. Γνωρίζω ότι από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση το παρέχουμε αυτό, θα το παρέχουμε αυτό, αλλά δεν ξέρω κάτι αντίστοιχο θα γίνεται από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το δεύτερο ερώτημα. Διαφάνεια και πώς είναι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Σας έδωσα το παράδειγμα του G-Cloud. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχει, δίνει τη δυνατότητα να, να συμπληρώσει τα στοιχεία που την αφορούν μια επιχείρηση μόνο μία φορά και όχι 20. Μόνο ε, επίσης τα στοιχεία που είναι συναφή για να γίνει ένα πρώτο screening, να γίνει μια πρώτη εξέταση του ποιε επιχειρήσεις μπορούν να ε, υποβάλουν προσφορά. Μετά, δεν έχω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για τις εξαγωγές μικρομεσαίων προς τις ε, Ηνωμένε όμως νομίζω ότι οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι κατά 5 10% λιγότερες από την αντίστροφη κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων και από την TTIP γενικότερα. Αλλά δεν έχω συγκεκριμένα αριθμιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ κύριος. Δεν είναι τόσο δύσκολο κανείς να βοηθά το εμπόριο στην αγορά. Ε, τι να κάνουμε, εγώ μόνος Αμερικανός και δεν είναι τόσο δύσκολο, επαναλαμβάνω. Εκεί που μένω εγώ είναι 100.000 ε, είναι αυτοί και περισσότεροι ε, είναι υπέρ αυτού και το ίδιο ισχύει και στο Υπουργείο Αμήνης και όσον αφορά ε, τα μαχητικά αεροπλάνα είναι ένα παράδειγμα συνεργαζόμαστε με Γαλλία και Γερμανία και βλέπετε ότι εκεί ζυγίζουν ε, το τι προσφέρουν οι ξένοι ε, και τι γίνεται με τους ντόπιου προμηθευτές. Για την Σλοβακία είπαμε ότι είναι από τις, ε, έχει από τους πιο διαφάνους διαγωνισμούς στον κόσμο και σε εμά σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχουμε αρκετή διαφάνεια. Ένας τομέας που είχε το πρόβλημα ήταν η συμφωνίε πλαίσιο. Οπότε στόχο μας για τα επόμενα χρόνια είναι ε, σε αυτού του είδους τις συμβάσεις πλαίσιο να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Και μιλάμε για 200-300 δις που καλύπτονται από τέτοιες ε, συμβάσεις. Τώρα σε επίπεδο πολιτιών και σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβάλλουμε περισσότερη ε, διαφάνεια. Τι μισούν την Ουάσινγκτον οι ντόπιοι. Και εγώ ο ίδιος άμα πάω σε κάποιον κυβερνήτη πολιτείας και του πω να έχει περισσότερη διαφάνεια μάλλον θα με κλείσει μέσα. Υπάρχει μεγάλη μεγάλη απέκτεια για την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οπότε υπάρχουν οι ομοσπονδιακές ενισχύσεις για να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα Και είπαμε, θα δούμε τα παλιότερα νομοθετήματά μας αν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε ή να τα καταργήσουμε. Και υπάρχει μεγάλη σιώδης οικονομία. Ας πούμε υπάρχουν ε, σε τοπικό επίπεδο και επίπεδο πολιτείας ε, ολόκληρη βιομηχανία πληροφορικής με κύκλους εργασίας κάποια δισεκατομμύρια ρωτήσατε γιατί ενώ θέλουμε ελεύθερη οικονομία, γιατί έχουμε την ε, προστατευτική νομοθεσία. Είναι ψυχολογικό αυτό. Είναι και πολιτική η λόγη. Ε, παίρνω το τρένο μεταξύ Νέας Υόρκης και Ουάσινγκτον και το τρένο αυτό που παίρνω κατασκευάστηκε το 78. Βγαίνω από εκεί με πονάει μέση μου. Οπότε εάν υπήρχε μια ευρωπαϊκή λύση ο κόσμος θα την ασπαζόταν αλλά δεν ξέρουν οπότε για αυτές τις προϋποθέσεις είπαμε σε τοπικό επίπεδο και επίπεδο πολιτείας ε, έχουμε έναν ε, πάρα πολύ αυστηρό νόμο κατά της ε, απάτης οπότε για τη διαφθορά και την απάτη θα ωφελούσε και σε αυτή την περίπτωση επομένω η συνεργασία. Θα σταθώ σε δύο στοιχεία που είναι τα πιο ενδιαφέροντα για μένα για το ζήτημα τη διαφθορά και τη διαφάνεια. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στι ΗΠΑ όπω και παντού. Οποτεδήποτε υπάρχει μια δημόσια σύμβαση μπορεί να υπάρξει ε, διαφθορά. Πολύ συχνά επίση γίνεται ε, στήσιμο των προσφορών, συμφωνούν μεταξύ του οι προσφέροντες. ή αξιοποιούν εσωτερική πληροφόρηση από την αναθέτουσα αρχή. Ο τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα είναι η διαφάνεια, είναι το ηλεκτρονικό σύστημα προσφορών, όταν αυτά τα στοιχεία είναι δημοσίω διαθέσιμα, περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια τη αναθέτουσα αρχή και μπορεί να αντιμετωπιστουν αυτα τα ζητηματα ειναι η διαφανεια ειναι το ηλεκτρονικο συστημα προσφορων οταν αυτα τα στοιχεια ειναι δημοσιω διαθεσιμα περιοριζεται η διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης και μπορει να γινει μεγαλύτερη διαφάνεια ανάθεση τελικά. Ε, γνωρίζουμε ότι στις, στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κριτήρια είναι πιο ξεκάθαρα και όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των υπαλλήλων κτλ. Πάντω θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στον τομέα τη διαφάνεια και, χωρίς την, και, και ανεξαρτήτω από την όποια συμφωνία με τι ΗΠΑ. Ο πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ε, παρουσιάσει θα τι βρείτε στην ιστοσελίδα της, των Επιτροπών ΙΜΚΟ και ΙΝΤΕ. Και θα ήθελα να ζητήσω ε, από τον εκπρόσωπο των συνδικάτων και από την κυρία Ντεχρούτ να μας δώσουν και εκείνη τις ομιλίες τους για να τις συμπεριλάβουμε στην ιστοσελίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα στους επόμενους ομιλητές και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σλέγγελμιχ, ο, ο οποίος είναι ε, Γενικό Διευθυντή και Διευθύνση Εμπορίου για τα ζητήματα επενδύσεων, πνευματική ιδιοκτησία και δημοσίων συμβάσεων. Επομένως καταλαβαίνετε πόσα δύσκολα θέματα έχει να αντιμετωπίσει. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά ε, του ε, συνδιοργανωτέ ε, τη ακρόαση. Είναι πραγματικά συναρπαστικό αυτό το αντικείμενο, όπω φάνηκε και από τι παρουσιάσει. Να σα δώσω και τι Διαστάσει από πλευρά των διαπραγματευτών του TTIP. Να προσπαθήσω να σας βάλω σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, να σας πω ποιε είναι οι τρει βασικές προκλήσεις για την πρόσβαση στην αγορά. Το επίπεδο της κρατικής ε, παρέμβαση και να σα μιλήσω και για κάποιου από τους κανόνες. Και μετά να απαντήσω και κάποια ερωτήματα. Καταρχά να σα πω ότι το θέμα της ε, συζήτησης για τις δυνατότητες δημοσίων συμβάσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ δεν είναι καθόλου καινούργιο Το συζητάμε 20 χρόνια τώρα και βάλε με τις είπα, για το πώς θα αυξήσουμε τις ευκαιρίες στην αγορές αυτές. Κάποιοι μιλήσατε για 12-15% του ΑΕΠ ή το μέγεθος της αγοράς πάντα συζητιέται. Γιατί αλλάζει, υπάρχει και διδικοποίηση, αλλά όπως και να το υπολογίσουμε είναι τεράστιο το ποσοστό αυτό. Είναι τεράστιο και Θέλουμε οικονομίε κλίμακα, θέλουμε σωστή δαπάνη του δημοσίου χρήματο και θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Δεν είναι μυστικό επίση ότι υπάρχουν πιο, πολύ, ε, πιο πολλά εμπόδια από αμερικανική πλευρά από τη ευρωπαϊκή πλευρά. Και στι διαπραγματεύσει, λοιπόν, ε, θα πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε αναγνωρίζοντα ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Γιατί στην αρχή υπήρχε σαφή στόχο του στόχου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες ε, για τις ε, επιχειρήσεις για να υπάρχουν μεγαλύτερες ε, ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση σε, σε ό,τι αφορά την εθνική αντιμετώπιση. Να μην υπάρχει δηλαδή διακρατική μεταχείριση και μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Πρώτη πρόκληση λοιπόν, να κοιτάξουμε την πρόσβαση στην αγορά. Προφανώς αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ που παραμένει το Buy American Act, πώς ε, δυσκολεύει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κτλ. Ένα επιχείρημα είναι ότι τελικά στην Ευρώπη παίρνουμε τελικά τα τις συμβάσεις αυτές για παράδειγμα, αναφέρθηκε το... αυτό που στην Ελλάδα το γεγονό ότι μα δυσκολεύουν πάρα πολύ μέχρι να πάρουμε τι συμβάσει αυτέ. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ε, Californian Railway Contracts. Πόσα ε, στοιχεία, πόσοι φορεί εμπλέκονται ε, για αυτό τι σημαίνει ότι η αλυσίδα παραγωγή θα πρέπει να προσαρμόζεται στου κανόνε αυτού ή ότι θα πρέπει να περνάμε δύσκολε να περάμε δύσκολε εξαιρέσει και πραγματικά είναι πολύ επίπονη η διαδικασία αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακόμα και αν ε, καταφέρουμε να πάρουμε συμβάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα εμπόδια αυτά, οι φραγμοί αυτοί. Και υπάρχει πραγματικά μεγάλη διαφορά. Κάτι που δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα. Το θέμα των set-asides που έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θα ξέρετε ότι 23% των ομοσπονδιακών συμβάσεων αυτόματα πηγαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ΕΠΑ με την λογική της υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Κατά πόσον όμως υπάρχει η ανάγκη να γίνει ε, τέτοια εξαίρεση και να εξαιρούνται οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες ε, επιχειρήσει σε ό,τι αφορά το θέμα των απευθεία αναθέσεων σε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και αυτό λοιπόν έχει το ρόλο του. Τελευταίο στοιχείο, αυξητική τάση. Δεν είναι παλιά αυτή η ιδέα του 19ου αιώνα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει νέα νομοθεσία η οποία ανακύπτει σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κυρίως από το Κογκρέσο, αλλά και από την Αμερικανική κυβέρνηση. Και υπάρχουν και οι πολιτείες ε, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, πριν από δύο χρόνια, επειδή από εβδομάδε καταφέραμε να του πείσουμε να πείσουμε τον κυβερνήτη τη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος, και στο Νέο Τζέρσι, να μην υπάρχουν στο Νιου Τζέρσι, να μην υπάρξουν, να μην μπουν καινούργιοι κανόνε. Σε ό,τι αφορά την Αμερική και σε ό,τι αφορά τις τοπικέ προτιμήσει. Αυτή είναι η βασική πρόκληση και είναι η πρόκληση που υπάρχει σε επίπεδο πολιτιών. Το δεύτερο βασικό θέμα στην διαπραγματεύσεις είναι τι θα κάνουμε σε επίπεδο πολιτιών. Γιατί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει απλά προδιαγραφές στις πολιτείες αυτό διαφέρει από τη, με την Ευρώπη, σε σχέση με την Ευρώπη, όπου συζητάμε, για παράδειγμα, σε κάθε κοινότητα να εφαρμόζει τις δύο, τις ίδιες, τις Υπάρχουν λοιπόν 7 πολιτείες που ε, έχουν ε, παρουσιάσει ζητήματα σε ό,τι αφορά και τον, τις προδιαγραφές του ΠΟΕ θέματα όπως για παράδειγμα τα συνεργατικές, συνεργατικές συμβάσεις πολίσεων δεν καλύπτονται για παράδειγμα από τις σχετικές προδιαγραφές. Το βασικό σημείο, μάλλον δύο βασικά σημεία και συνδέεται αυτό με το τρίτο θέμα των κανόνων. Καταρχάς δεν υπάρχουν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σε ό,τι συμβαίνει σε επίπεδο πολιτείας. Δεν υπάρχει ε, τρόπο τρόπος ε, αναφοράς, δεν υπάρχει κεντρική ε, βάση δεδομένων όπως στην Ευρώπη. Άρα ένας στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε ακριβώς στο σημείο αυτό. Αντιθέτως από την εντύπωση που δίδεται, αυτό το θέμα για τη διαφάνεια είναι βασικό θέμα των διαπραγματεύσεων. Προτείναμε να υπάρξει η μια κεντρική βάση δεδομένων, ένα κεντρικό κόμβο όπου θα μπορεί κανεί να βρίσκει όλε τι δημόσιε συμβάσει σε επίπεδο ΙΠΑ, όπω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φυσικά τίθεται μετά και το θέμα του κατά πόσον μπορεί να κάνει κάποιο καταγγελία, κατά πόσον μπορεί μια ε, επιχείρηση να συμμετάσχει. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα προς τις πολιτείες πέρα από το κατά πόσον δεσμεύονται ότι ήταν ανοιχτές και διαφανείς ε, οι διαδικασίες ε, για τις δημόσιες προμήθειες υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας. Αλλά φυσικά χρησιμοποιούν πολύ ομοσπονδιακή χρηματοδότηση οι πολιτείες ε, και οι πολιτείες λοιπόν όταν εκτελούν μεγάλα έργα υποδομών πολύ συχνά χρησιμοποιούν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για την υδροδότηση, είτε πρόκειται για άλλα ζητήματα. Και μπορεί λοιπόν να κάνει κάτι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δεν μπορούν να προδιαγράψουν του κανόνε για τι δημόσιε προμήθειε, αλλά μπορούν να βάλουν αιρεσιμότητα στα κονδύλια που δίδονται. Να του πει, για παράδειγμα, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν προτιμήσει όταν χρησιμοποιούνται ομοσπονδιακοί πόροι. Και αυτό απαντάει και σε κάποιες από τις προτάσεις. Το έχουμε εξετάσει το ζήτημα αυτό και θα θεωρούσαμε ότι θα ήταν μεγάλο επίτευγμα αν οι ομοσπονδιακοί κανόνες απλά θα προδιάγραφαν, προδιάγραφαν ότι δεν ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, οι ομοσπονδιακοί πόροι, αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή επιδοτήσεων. Τρίτο ζήτημα για τους κανόνες. Σε ό,τι αφορά και το θέμα και της διακυβέρνησης και της διαχείρισης, το με αυτό το θέμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί πρόκειται για το θέμα ε, των ε, χρημάτων, των φορολογουμένων, των ε, κατανάλωτων, γιατί πρόκειται για πολύ μη αποδοτικό και χρονοβόρο και δαπανηρό τρόπο διεξαγωγής των δημοσίων συμβάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέτουμε το θέμα των κοινωνικών ή πράσινων προδιαγραφών στις δημόσιες προμήθειες. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το υποστηρίξουμε, γιατί όσον δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, μιλάμε για διακριτική μεταχείριση, δεν μιλάμε για άλλους στόχους όπως η οικολογική επισήμανση. Εδώ είμαστε ανεκτοί, γιατί δεν θεωρούμε ότι το άνοιγμα των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να αγγίζει τους στόχους αυτούς και τα θέματα αυτά. Θέλουμε να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα ανοιχτή αγορά. Όχι να τύφονται στόχοι τέτοιοι για την οικολογική επισήμανση. Αυτό το προωθούμε με, μέσω άλλων τομέων. Να προσπαθήσω να απαντήσω και κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαι σύντομο, αν μου το επιτρέπετε, γιατί δεν έχω και χρόνο. Το θέμα, ε, για παράδειγμα, της ε, παράκαμψης μέσω Καναδά ετέθησε. Και το ίδιο ισχύει και για την Ελβετία και για άλλες χώρες, ότι αν έχει κανείς έδρα εκεί μπορεί να κάνει κανείς ε, μια κοινή επιχείρηση, αλλά ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, γιατί το θέμα δεν είναι που είναι η έδρα στην Καναδά ή σε ΣΥΠΑ, αλλά ποιες υπηρεσίες παρέχονται. Το να διοικητεύσουμε λοιπόν ε, τις υπηρεσίες και τα αγαθά μέσω Καναδά δεν ε, αλλάζει τίποτα αν δεν αλλάξουν οι κανόνες της προέλευσης. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας λοιπόν ετέθησε και το θέμα του καμποτάζ. Και πάλι, εδώ θεωρώ ότι πρόκειται για τεχνική λεπτομέρεια. Το καμποτάζ είναι και προβλέπει το ποιο παρέχει την υπηρεσία, αλλά όχι το πιο πλοίο, σε ποιο πλοίο παρέχει ο πάροχο την υπηρεσία. Μια μεγάλη διαφορά λοιπόν είναι το καμποτάζ μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι ανοιχτό από πλευρά των ΗΠΑ. Η κατάσταση είναι συγκρίσιμη. Δεν υπάρχει μεγάλο καμποτάσταση στην Ευρώπη γιατί δεν είναι μεγάλε οι αποστάσει. Αλλά εδώ πέρα, σε ό,τι αφορά του κανόνε ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, από τα παραδείγματα που έχουμε, το θέμα δεν είναι κατά πόσο μπορεί να παρέχει κανεί την υπηρεσία. Αλλά οι επιχειρήσει που, που αγοράζουν, για παράδειγμα, παγοφλαστικά φέρει σε, σε, με δημόσια ε, ιδιότητα, τι τίθεται το θέμα του κατά πόσον το πλοίο θα πρέπει να είναι αμερικανικό ή όχι. Το οποίο ό,τι αφορά τι δημόσιε υπηρεσίε αποτελεί πρόβλημα. Ένα θέμα που έθεσε ο κ. Κασπάρη για τι ε, δημόσιε ε, και κοινοφιλέ υπηρεσίες. Συμφωνώ και επαυξάνω. Όταν μιλάμε για δημόσιε συμβάσει δεν κοιτάμε το, το τι υπηρεσία ε, παρέχει το κράτος στην ελεύθερη αγορά και όλα αυτά δεν σχετίζονται. Οι κοινοφελεί υπηρεσίε δεν σχετίζονται. Δεν πρόκειται να τα αλλάξουμε αυτά. Δεν, πρόκειται να... δεν προσπαθούμε καν να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία. Υπάρχουν λοιπόν δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν δήμοι κοινότητες οι οποίες δεν καλύπτονται πολύ απλά. Ο βασικός μας κανονισμός για τις δημόσιες συμβάσεις δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Ένα άλλο ερώτημα του κυρίου Κασπάρη για το μέγεθο των ευκαιριών και των δυνατοτήτων. Και εδώ περνάμε σε επίπεδο στατιστική, ε, το οποίο το συζητάμε συχνά και με του Αμερικανού ομολόγου μα. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Κανεί δεν αναφέρει αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να ξέρουμε τον αριθμό των συμβάσεων, αλλά από, πού προέρχονται τα αγαθά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσουμε. Πόσο μάλλον και με τι σύγχρονε αλυσίδε ε, παροχή. Έχουμε κάποιες, ε, κάποια αριθμητικά στοιχεία που υπολογίζουμε, το αμφισβητούν οι Αμερικανοί, αλλά δεν είναι επιστημονικά αυτά τα στοιχεία. Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία, πολύ ομαδοποιημένα όμως από πλευρά ε, των ΙΠΑ και έχουμε και κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποιες εικασίες. Αλλά επικεντρωθούμε στα βασικά εμπόδια. Γιατί αν ρωτήσουμε τις επιχειρήσεις ποια είναι τα προβλήματά τους, δεν θα μας μιλήσουν για τα στατιστικά στοιχεία, μας λένε ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Δύο άλλα στοιχεία. Απαντώντα στα ερωτήματα του κ. Βίνκλερ και άλλων, αναφερθήκατε στη ΣΥΤΑ. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα της, ε, των θεωρήσεων. πάντοτε θέτουμε το θέμα, ε, το έχουμε θέσει και στον Καναδά, να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα ε, με τα κράτη-μέλη για τα οποία ζητούνται ε, θεωρήσεις ακόμα. Νομίζω υπάρχει και ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο δεν απάντησα, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι. Μπορείτε να μου το θυμίσετε. είναι περισσότερο ζήτημα εμπορίου. Είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το παρακολουθεί. Για το, την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις λοιπόν. Ε, πράγματι, οποτεδήποτε μια οδηγία είναι περίπλοκη, τίθεται το θέμα του πότε θα τεθεί σε εφαρμογή και αν θα γίνεται αυτό σωστά. Δεν ξέρω όμως πιο συγκεκριμένα να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε με τους μάλλον θα σας, ευχηθώ καλή τύχη στον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων, στο 13ο. Και έχουμε φτάσει στο τέλος της συνάντησης μας. Έχει την δυνατότητα ντίτα ως ε, η συγγήτρια από την πλευρά της ΙΜΚΟ να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί με τις κυριότερες πτυχές της διαπραγματεύσης ε, της TTIP. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, ιδέες και απόψεις για το τι θα μπορούσαμε να θέσουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και εγώ ένα από τα συμπεράσματα που κρατώ είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ποιους θέλουμε να ωφελήσει αυτή η συμφωνία και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι από τις ωφελούμενες. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσουν τους ομολόγους τους από τις ΗΠΑ ε, γιατί γνωρίζουμε ότι και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι, οι πιο, είναι η της οικονομίας, είναι εκείνες που δίνουν τις μεγαλύτερες, τις περισσότερες θέσεις εργασίας και καινοτομούν. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θέλουμε να κινηθούμε στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και εδώ νομίζω συμφωνούμε ότι σε όλα τα επίπεδα οργάνωση του κράτους. Θέλουμε να υπάρξει άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων και στο ε, ομοσπονδιακό και στο πολιτιακό και στο τοπικό ευελπιστώ οι διαπραγματευτές μας να καταφέρουν να πείσουν τους ομολόγους τους να διαγραφτούν αυτές οι τρεις λέξεις από την νομοθεσία που μας ανέφερε ο κ. Καθηγητής που θα δώσουν την δυνατότητα να ανοίξουν οι δημόσιες συμβάσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους στόχους εδώ, στον αφορά δηλαδή τις δημόσιες συμβάσεις και νομίζω ότι αν το καταφέρουμε θα βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στην αμερικανική αγορά. Και θα σα μιλήσω σαν εισηγητή για το Κοινοβούλιο τη Διατλαντική Συμφωνία. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ του ε, ομιλητέ μα. Νομίζω ότι μα βοήθησαν σήμερα το πρωί γιατί μα μίλησαν για ε, αυτά τα τόσο δύσκολα θέματα τα πιο δύσκολα των ε, διαπραγματεύσεων και κατά τη γνώμη μου αυτό θα, θα, μπορούσε τώρα να είναι η αρχή μιας καινούργιας φάσης γιατί έχουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα συζητούμε δημοσία αλλά αυτό το οποίο σήμερα συζητήσαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις διαπραγματεύσεις που καλά κρατούν εδώ και τρία χρόνια χωρίς να υπάρχει τη σήμερα ημέρα κάποια πρόοδος. Και αν στον επόμενο γύρο δεν έχουμε πρόοδο και στους επόμενους δύο γύρους, τότε τον Ιούλιο θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε εάν θέλουμε να συνεχίσουμε ή εάν θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι σύντομα δεν μπορεί να κλειστεί μια συμφωνία. Βεβαίως και τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχουν ένα σωρό εμπόδια ακούσαμε σήμερα το πρωί και ήδη όσον αφορά τα διάφορα επίπεδα, όπως είπε η Ντίτα, το ομοσπονδιακό, το υποομοσπονδιακό επίπεδο, τη χρηματοδότηση ε, που προέρχεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και σε υποομοσπονδιακό επίπεδο, τους κακούς που μπλέκονται. Άρα θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας και στατιστικά στοιχεία γιατί ε, βλέπουμε ότι και όσον αφορά τις προμήθειες υπάρχουν ε, διάφορα μέτωπα ε, και δημοσιονομικά και φορολογικά και κοινωνική πολιτική και όλα αυτά θα πρέπει να τα χειριστούμε με συνέπεια, με λογική και να προσφέρουμε κάποια αποτελέσματα θετικά για τις ΜΜΕ αλλά και για τους ε, αλλά και τους εργοδότες. Άρα θα πρέπει να προκύψει ένα αποτέλεσμα θετικό για όλους. Παρ' αυτά, τα πράγματα επιδέχονται βελτίωση από ευρωπαϊκής πλευράς. Είμαι αισιόδοξος. και ελπίζω οι διαπραγματευτές θα μπορέσουν να προχωρήσουν και τον Ιούλιο να μην θεωρήσουμε ότι φτάσουν στο τέλος της διαδρομής. Και πάλι πρέπει να ευχηθούμε καλή τύχη στους διαπραγματευτές για τον επόμενο γύρο. Φόρντ. Και εγώ να ε, δευτερολογήσω και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο για την Επιτροπή Ιστορική Αγορά στο κεφάλαιο των προμηθειών και γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει να βοηθήσουμε τις διαπραγματεύσεις γιατί για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς υπάρχουν πολύ θετικές δυνατότητες και το μήνυμα που πήρα ήταν πολύ θετικό από την Ομοσπονδία των Μικρών Επιχειρήσεων. φαίνεται ε, πάρα πολύ θετικό να υπάρξει διαφάνεια και κάποιες πρακτικές ιδέες από το δεύτερο πάνελ για το πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία στα ψηφιακά και πώς μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις ούτως ώστε να διευκολυνθεί η υπόθεση των ε, προμηθειών δυνάμει της συμφωνίας TTIP. Όλοι βέβαια θέλουμε να βοηθήσουμε ε, τις ε, τοπικές επιχειρήσεις Α, και ακούσαμε κάποιες πρακτικές ιδέες και συμφωνώ με την Τίτα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε να μην πούμε ότι εδώ είναι το τρόπο της διαδρομής να βρούμε πρακτικές λύσεις για να διευκολύνουμε την υπόθεση των ε, προμηθειών και δύο σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως τα ψηφιακά ξέρουμε ότι πρέπει και σε διεθνέ επίπεδο και όχι μόνο στην Ευρώπη να προσπαθούμε να αφήσουμε όλες τις πόρτες ανοιχτές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε θα ωφεληθούν όλοι και οι δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Επίση πρέπει να σας πω ότι εκεί δίπλα στην είσοδο της αίθουσα έχουμε αυτά τα φυλάδια σε σχέση με τις ευρωπαϊκέ ρυθμίσει για τι προμήθειε. και ίσως ε, μπορούν, θέλετε αυτά να τα πάρετε και να τα προωθήσετε στους ε, περιφερειακούς οργανισμούς σας γιατί αυτά είναι πρακτικά για τον κόσμο που ασχολείται με το θέμα και εγώ το έχω κάνει αυτό. Αυτά τα φυλάδια είναι, λέει η κυρία Φόρτ και τα δείχνει, υπάρχουν και στην, κοντά στην είσοδο και θα δείτε πώς λειτουργεί η πολιτική προμηθειών της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας ευχαριστώ ευχαριστούμε και για την αγαστή συνεργασία των Επιτροπών μας. Και εγώ ευχαριστώ για τη συνεργασία. Σε δύο λεπτά θα αρχίσει η, η συνεργασία, η, συγγνώμη, η συνεδρίασή μας στο 1, η Επιτροπή μας, συγγνώμη, στο 1α σε αυτό το κτίριο, 1α002.